σας υποβάλει ερώτηση. Συμφωνείτε, κύριος Μπρέαρ. Αγαπητέ συνάδελφε, από εδώ, είπατε ότι δεν θέλετε να χάσει την νομοποίηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζετε την ιδέα του θεμελιώδους ε, κοινωνικού συμβολέου του Ρωσό και ότι οι πολίτε θα πρέπει να συμφωνούν για το τι είδου κυβέρνηση θέλουν. Θεωρείτε ότι αυτή η ιδέα απειλεί την αντιπροσωπευτικού τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς ή μήπω συμφωνείτε ότι έχουμε εκλεγεί για να εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Συγγνώμη, αλλά έχει περάσει ο χρόνος σας. Υπάρχει και δεύτερη ερώτηση με την μπλε κάρτα. Κύριε Γκοσάλες Πόνς, παρακαλώ. Έστεμπαν. Και άλλο συνάδελφο έχει ζητήσει ε, με μπλε κάρτα το δικαίωμα να υποβάλει ερώτηση. Εγώ πιστεύω στην αντιπροσωπευτική εντολή, στη βουλευτική αντιπροσωπευτική εντολή. Αντιλαμβάνομαι ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλουν διαβουλεύσει με του πολίτε, γιατί δεν είναι κοινοβούλια το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ όμω ότι υπάρχει μία αντίφαση μεταξύ όσων. Υπάρχει μια αντίφαση. Ε, Ευρωβουλευτέ, οι βουλευτέ που έχουν εκλεγεί πολύ πρόσφατα, πριν από έξι μήνε από του πολίτε, να πρέπει να ξαναδιαβουλευτούν με του Ευρωπαίου πολίτε. Συγγνώμη, αλλά μισό λεπτό είχα, δεν μπορούσα να επεκταθώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ενδιαφέρονται όλα αυτά. Συγγνώμη, δεν ξέρω το μικρό σας. Και άλλοι περιμένουν να μιλήσουν, οπότε θα περάσουμε στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Ρουίς Δεβέσα, γιατί αρχίζουμε και μένουμε πίσω στο χρόνο. Δεν θα δεχτώ την 92η ώρα της μπλε κάρτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω στους συναδέλφους από την άκρα δεξιά ότι έρχονται κάθε μέρα εδώ στο Κοινοβούλιο για να μας πούν τι σκέφτονται, τι πιστεύουν και τι νιώθουν οι πολίτες και θεωρούν ότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε λάθος. Εσείς όμως εκπροσωπείτε μόνο 20-25% των Ευρωπαίων πολιτών. Οι φιλευρωπαϊκές ομάδες που εκπροσωπούν πάνω από 75% των Ευρωπαίων πολιτών συνέταξαν το σχετικό ψήφισμα. Οπότε Ας δούμε εδώ πώς έχει κατάσταση και πόσοι εκπροσωπούν ποιους. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τη θέση ισχύ της ηθίκης της Λισαβόνας και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ο κόσμος σήμερα έχει αλλάξει ριζικά από τον κόσμο το 2009. Τότε δεν είχαμε ούτε Brexit, ούτε Αραβική Άνοιξη, ούτε τον Τραμπ, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είχαμε μεταναστευτικές ροές τότε. Οπότε, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους που αναφέρθηκαν ε, το Φρόιντ ε, και τις ε, ουσίες που μας συναρκώνουν. Όχι, δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα, τη βλέπουμε πολύ καλά, βλέπουμε τις εξωτερικές πιέσεις και θα πρέπει να αντιδράσουμε. Και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να μας καθοδηγήσει, γιατί ο κόσμος είναι εκεί, δεν μπορούμε να τον αγνοούμε θα πρέπει να μα οδηγήσει σε μια πολιτική ένωση φεντεραλιστικού τύπου. Αυτό όμω θα το κάνουμε από κοινού με τους πολίτες, σε συζητήσει με του πολίτε και με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε και τη συμμετοχή τη Οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Πιστεύω ότι μπορούμε ε, να εμπλέξουμε και τους πολίτες και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στη διαδικασία και τους εθνικούς βουλευτές και στη συνέχεια να καταλήξουμε σε μια σειρά απαντήσεων στις προκλήσεις πολιτικής που αντιμετωπίζουμε και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Και έτσι μπορούμε ε, να αντιληφθούμε τις προκλήσεις, να δώσουμε και τις σωστές θεσμικές απαντήσεις. Υπάρχει μια ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Τη δέχεστε? Τη δέχεστε κύριε Ντεβέσα? Ναι. Μισό λεπτό. Ο κύριος Ζόντσα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον συνάδελφο. Το 1992 εγκρίθηκε η συνθήκη του Μάστριχτ που προέβλεπε την Ένωση των Πολιτών. Ήδη από το 72. Ε, από το 92, συγγνώμη, τη συνθήκη του Μάστριχτ. Γιατί λοιπόν δεν τα καταφέραμε, γιατί τόσα χρόνια έχουν περάσει και δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο που προβλεπόταν ήδη από τη συνθήκη του Μάστριχτ του 92. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά την ερώτηση. Την πολιτική ένωση, τι σημαίνει, ένωση των πολιτών, τι εννοούσατε ακριβώς. Καλώ τότε να τα βρείτε ε, διμερώς αργότερα. Η κυρία στο έδρανο 29 ζήτησε επίσης ε, με την μπλε κάρτα ερώτηση. Ευχαριστώ. Απολαμβάνω την ε, συζήτηση αυτή και χαίρομαι που έχουμε τις μπλε κάρτες γιατί για πρώτη φορά νιώθω ότι έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση που είναι απαραίτητη όταν μιλούμε για το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρίες να δώσω λίγο από το χρόνο μου στον συνάδελφο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, που μίλησε για την ανάμειξη των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο μέλλον της Ευρώπης και στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό θα ζήτησα το λόγο με την μπλε κάρτα, για να του δώσω λίγο ακόμη χρόνο να μας αναπτύξει αυτή την πρότασή του για την ανάμειξη στη διαδικασία και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τη κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω, πιστεύω στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως και ο συνάδελφος Γκοσάλες Πόνς, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία αντίφαση μεταξύ της, αντιπροσωπ... της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της μόνιμης διαβούλευσης με τους πολίτες. Είμαστε αιρετοί ε, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει καθημερινά να έχουμε επαφέ με του απλού πολίτε, με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και θα πρέπει να το κάνουμε και στα πλαίσια τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε αιτήματα 16 ήδη αγορητών για τη διαδικασία Catch the Eye. Επομένω, θα κλείσω τον κατάλογο, αλλά θα κρατήσω τις μπλε κάρτε. Για δύο λεπτά η κυρία Ντυρόν θα είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ο κύριος Ντυρόν, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ακούσατε τη θέση του Κοινοβουλίου, η οποία είναι σχεδόν ομόφωνη, όσον αφορά την ανάγκη να επιτύχει αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο εγγράφεται σε μια συζήτηση που μερικές φορές είναι υπερβολικά ε, θεσμοθετημένη. Ε, χρησιμοποίησατε μια λέξη, κυρία Συνέλφη, προηγουμένως. Ε, αναφερθήκατε στην λέξη τόλμη Ξέρετε ότι ο επαναστάτης Νταντών ε, είχε αναφερθεί στη φράση αυτή λέγοντας ότι χρειαζόμαστε τόλμη, ξανά τόλμη, περισσότερη τόλμη, πάντα τόλμη. Του λοντάς στα γαλλικά. Ε, βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Χτες συζητήσαμε για το Brexit, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα και άλλοι κίνδυνοι. Ε, στην ε, ε, πλατεία Κλεμπέρ εδώ στο Στρασβούργο στο τέλος του πολέμου ο Σούμαν έλεγε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη η οποία θα, είναι, θα αντλεί την δύναμή της από την ενότητά της θα βασιστώ σε μια φράση του Ζαμονέ. Ο Ζαμονέ έλεγε όταν δημιουργήθηκε η Ευρώπη ότι η Ευρώπη δεν είναι εδώ για να συνασπίσει χώρες, ε, είναι εδώ για να συνδέσει τα ε, άτομα, τους πολίτες, τα ανθρώπινα όντα μεταξύ τους. Ε, αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Στρέφομαι λοιπόν προς το Συμβούλιο με ανησυχία ε, και με ελπίδα όμως. Στρέφομαι και προς εσάς ε, κυρία Σουίτσα και προς το Συμβούλιο και προς την Κομισιόν στρέφομαι έτσι ώστε ε, να σας ζητήσω εξ ονόματος των μη κυβερνητικών οργανώσεων που χτυπούν την πόρτα των θεσμικών οργάνων. Σας ζητώ εξ ονόματος της κοινωνίας των πολιτών να μην χαλάσετε, να μην σπαταλίσετε αυτή την ευκαιρία που έχουμε για να δουλέψουμε όλοι μαζί, το σύνολο όλων όσοι εκπροσωπούν τους ε, πολίτες και την οργανωμένη ζωή των πολιτών. Όλοι μαζί, γιατί δεν μπορούμε να επιτύχουμε οι μεν χωρίς τους δε. Ζητήσατε catch the eye ή μπλε κάρτα, παρακαλώ, αγαπητέ συνάδελφε. Ωραία. Ε, μία ερώτηση με μπλε κάρτα από τον κύριο Καστάλντο. Τι δέχεστε κύριε Ντυρό. Ναι. 30 δευτερόλεπτα έχετε διάθεση. Αγαπητές συνάδελφε, α, ε, πολύ αγαπημένα μου Πασκάλ, έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια σε πολλά σημαντικά θέματα. Ε, είδαμε ότι προσδοκούμε από την διάσκεψη ε, ε, πολλά πράγματα, αλλά ίσως δεν θα οδηγήσει σε μεταρρύθμιση των συνθήκων. Δεν θεωρείται όμως όπως και εγώ ότι θα πρέπει να έχουμε και σαν ενδεχόμενο την διάσκεψη των ε, συνθήκων στα πλαίσια αυτής της διάσκεψης έτσι ώστε να επαναισορροπηθούν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι πολύ ισορροπημένα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Φάμπιο νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά αυτά που είπε το Συμβούλιο και η κυρία Σουίτσα από την Κομισιόν. Ε, δεν πρέπει να προδικάσουμε τίποτα, δεν πρέπει να απαγορεύσουμε στους εαυτούς μας, αυτούς μας τίποτε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο που είναι απαραίτητος έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε λύσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εμπλοκές ε, στην Ευρώπη. Ας δείξουμε τόλμη να μην φοβόμαστε τους Ευρωπαίους πολίτες, να μην φοβόμαστε τον διάλογο και όντω να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε, να μεταρρυθμίσουμε ό,τι πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Για 1,5 λεπτό η επόμενη ομιλήτρια θα είναι η κυρία Ντελμπό Σκορφίλντ. Μελετούμε το κείμενο για την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, τον Ιανουάριο που όπως υπόθηκε και προηγουμένως είναι η τελευταία παρουσία των Βρετανών συναδέλφων. Ε, και θα έχουμε λοιπόν την αποχώρηση, του, της, την πρώτη αποχώρηση ε, μιας χώρας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η μόνη αποχώρηση. Επίσης ε, συζητήσαμε και ένα ε, ε, ψήφισμα για το άρθρο 7 και την ενεργοποίησή του εναντίον της Πολωνίας και της Ουγγαρίας για θέματα κράτους δικαίου. Φαίνεται ότι αυτές οι απειλές είναι σημαντικές, αλλά εμείς από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε την δυνατότητα να αντιδράσουμε. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι αξιοσημείωτη προσπάθεια και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και να αξιολογήσουμε θετικά την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που προσυπέγραψε αυτήν ε, την ε, διαδικασία. Αλλά δεν θα πρέπει να πλανόμεθα. Εάν αποτύχει η διάσκεψη θα είναι αποτυχία και για τα τρία θεσμικά όργανα και θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την απώλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπω τη θέλουμε, δηλαδή βιώσιμη, προοδευτική και συμπεριληπτική. Εμείς ε, εργαζόμαστε εδώ ως ε, Ευρωπαίοι βουλευτές ε, σε πολύ προνομιούχες συνθήκες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Γαλλία και στην Ιρλανδία και στη Γερμανία υπάρχουν πολίτες, άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν για μας πηγή έμπνευση. Θα πρέπει επομένως να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους αυτούς. Θα πρέπει να τους δώσουμε την τεχνογνωσία. Θα πρέπει να τους γραστούμε τις ανάγκες τους. Διακόπτει η Πρόεδρος στο μικρόφωνο της ομιλήτρια. Δεν υπάρχει λόγο να ξεπερνάτε το χρόνο σα, γιατί θα αναγκάζομαι να σα ε, ε, κλείνω το μικρόφωνο και δεν θα υπάρχει και συζήτηση. Ο διάλογο που κάνουμε τώρα. Σα παρακαλώ λοιπόν να μην το κάνετε. Ένα μισή λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Άνεμαν, συνάδελφοι. Ας μην ε, χρονοτριβούμε εδώ σήμερα. Αυτή η μεγάλη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είτε έχει ως σκοπό αυτή την αντίσταση των, ε, της καταπολέμησης της διάβρωσης της εθνικής επικυριαρχίας να σταματήσει και τα τελευταία χρόνια έχουμε την αίσθηση ότι αυτό είναι το αίσθημα το που ανακύπτει από όλε τι εκλογέ τα τελευταία χρόνια. Λιγότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο πολύ ελευθερία σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία ή είναι μια μορφή θεάτρου ε, τύπου Μακρόν για να παραμεριστούν τα πραγματικά προβλήματα. Πολύ φοβόμαστε αυτό το τελευταίο ισχύει γιατί στα τρία σημεία στο κείμενο εμφανίζεται τέτοια στοιχεία και παρά την αντίστασή μας η Αναφέρεται διαρκώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστεί μια πιο στενά συνεργαζόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένα θέατρο αυτό. Είναι ακριβή αυτή η παράσταση, είναι άχρηστη και δίνει όλο και πιο πολλέ αρμοδιότητε στην Ευρώπη αυτή. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Τι πρόεδρο, για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Μπουρζόν. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Συνάδελφοι, η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι δύο εκπρόσωποι των πολιτών είναι τα εθνικά κοινοβούλια και το κοινοβούλιο αυτό. Και είναι καλό να ακούμε τι λένε οι πολίτες, οι ΜΚΟ, αλλά ποτέ δεν είμαστε αντιπροσωπευτικοί. Αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι πολιτικούς, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίοι τολμούν να αποφασίσουν και οι οποίοι είναι υπόλογοι για τις αποφάσεις τους. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και θέλουμε να υπάρχει μια επιπρόσθετη αξία. Αν δεν υπάρχει επιπρόσθετη αξία, ας μείνουν τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Πιο πολύ ιστορική αγορά, πιο πολλά ε, συνοριακή διαφύλαξη των συνόρων, αλλά ας μείνουν τα εθνικά σε εθνική επιχειριαρχία. Ευχαριστώ, κύριε Φερέιρα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκείνοι που ε, κυβερνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν προσποιούνται ότι θα φουγκραστούν τους λόγους της Ευρώπης. Αυτό είναι όμως φάρσα, φαρσοκομωδία, γιατί ε, επιτρέπουν δημοψηφίσματα μόνο όταν τους βολεύουν, εφαρμόζουν λιτότητα, ενώ όταν ε, κάνουν δημοψηφίσματα που δεν τους αρέσουν ε, ε, υπαναχωρούν. Και τώρα τάχα θέλουν ευρύ ανάμειξη των Ευρωπαίων πολιτών για να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη φαρσοκομωδία. Υποτίθεται ότι δεν θα προδικάσετε τίποτα, δεν θα προεξοφλήσετε το αποτέλεσμα. Εμεί όμω είμαστε εδώ για να δώσουμε μάχη για νέα Ευρώπη, όχι την νεοφιλελεύθερη των πολυεθνικών ομάδων και εταιριών. Είμαστε κατά μια στρατιωτικοποιημένη Ευρώπη. Είμαστε μια Ευρώπη των πολιτών ε, και τη ειρήνη, όχι μια Ευρώπη ισχυρών. Είμαστε μια Ευρώπη ισότιμων κρατών και ισότιμων πολιτών. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την Ευρώπη και κυρίω βρισκόμαστε εδώ για να τη μεταρρυθμίσουμε, για να τη μεταμορφώσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πουτζδεμόν για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν διαρωτόμαστε για το μέλλον της Ευρώπης, το πρώτο που θα πρέπει να λύσουμε και να απαντήσουμε είναι τι ρόλο θα δώσουμε στους πολίτες. Αν δεν λύσουμε αυτό το θέμα, σε λίγα χρόνια θα επαναληφθεί η ίδια συζήτηση με άλλους ευρωβουλευτές και θα, ήταν, θα είναι δική μας αποτυχία. Θέλουμε η πολίτες να είναι απόμακροι και αδιάφοροι ή να μετράει πραγματικά η φωνή τους και η άποψή τους και να συμμετέχουν άμεσα, απευθεία στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Θέλουμε λοιπόν να επιτρέψουμε μηχανισμούς και να θεσπίσουμε μέσα για να συμμετέχουν οι πολίτες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία μας για να μην ρίχνουμε νερό στο μήλο των λαϊκιστών. Γιατί ε, εναλλακτική λύση δεν θα πρέπει να είναι ο πειρασμό των ευρωσκεπτικιστών. Η Ευρώπη δεν είναι για τους κομφορμιστές και τους σκεπτικιστές, αλλά για τους ε, απαιτητικού. Κύριε Πουσδεμόν, δέχεστε ερώτηση με μπλε κάρτα από την κυρία Μοσαράτ, βεβαίως. Έχετε το λόγο, κυρία Μοσαράτ. Η Ευρώπη είναι ένα πολιτικό σχέδιο ε, που στηρίζεται στο κράτος δικαίου και την ισχύ του νόμου. Είναι μια κοινότητα αξιών στην οποία συμμετέχει και η Ισπανία. Η Ευρώπη είναι το αντίδοτο στον καταστροφικό σας εθνικισμό. Ε, εσείς επιτεθήκατε ε, στο κράτος δικαίου και υπεξαιρέσατε δημόσια κονδύλια. Και τώρα φοβάστε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί ασυλία δεν σημαίνει ατιμορρησία. Κανεί, έστω και ευρωβουλευτή, δεν είναι περάνω του νόμου. Πότε θα έχετε το κουράγιο, πότε θα χάσετε το φόβο να αντιμετωπίσετε. Δυστυχώ κλείνει το μικρόφωνο τη ομιλήτρια. Έχετε το λόγο, κύριε Πουσδεμόν. Κυρία Μονσεράτ, νομίζω ότι εσεί θα πρέπει να σεβαστείτε του κανόνε που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει οδηγία που εμποδίζει τους δημόσιους αξιωματούχους ε, και τους ευρωβουλευτές ε, να μην χάνουν το, το τεκμήριο της αθωότητας. Σε τι καταδίκες αναφέρεστε, σε τι δίκες αναφέρεστε, σε τι εγκλήματα αναφέρεστε, τι εγκλήματα διέπραξα εγώ ε, για να με κατηγορείτε έτσι. Πιστεύω ότι οι χώρες θα πρέπει να τηρούν τους νόμους και το, η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υποστεί κυρώσεις γιατί ακριβώς παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σταγιάννη για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης είναι να επιστρέψουμε στην πολιτική. Η μεγάλη, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση είναι να έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές και εξωτερικές ε, προκλήσεις. Ε, βεβαίως χρειαζόμαστε Ευρώπη με ενιαία εξωτερική πολιτική, με ενιαία αμυντική πολιτική. Είδαμε ε, την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση της Συρίας, στην κρίση της Λιβύης, όσα συνέβησαν στην ε, Βενεζουέλα. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν συνεκτική και δυναμική δράση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ε, να ξεχάσουμε τις εθνικές ταυτότητες ή τα εθνικά κράτη. Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να ε, αποτελέσει το πρόσχημα για την καταστροφή των μικρών πατρίδων. Αντιθέτως η Ευρώπη υπάρχει έτσι ώστε να διευρύνει την έννοια της πατρίδας. Ούτε πιστεύω ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με δημοψηφίες ψηφίσματα νομιμοποιημένα ή όχι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε λύσεις μέσα από μια πραγματική δημοκρατία, όχι από ε, ε, μη ε, εκπροσωπευτική, αντιπροσωπευτική συγγνώμη, δημοκρατία η οποία θα αντιτίθεται στις θελήσεις τις εκπεφρασμένες άλλωστε των λαών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την νομοθετική πρωτοβουλία όπως γίνεται σε όλα τα κοινοβούλια. Βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε δώσουμε χώρο να ακουστεί η φωνή ε, των πολιτών, αλλά θα πρέπει να δώσουμε κυρίως ε, ε, χώρο να ακουστεί η φωνή των ερετών, των ήδη εκλεγμένων δημάρχων, περιφερειαρχών κλπ. Ευχαριστώ. Σίλβα Περέιρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα είναι καλή ευκαιρία για να ξαναέρθουν κοντά οι πολίτες στο ευρωπαϊκό σχέδιο, αρκεί να τηρηθούν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να έχουμε μια πραγματικά ανοιχτή συζήτηση ευρεία συμμετοχή, όπου όλοι οι πολίτες και οι αντιπροσωπευτικέ του οργανώσεις να μπορούν να εκφέρουν τη γνώμη τους και να ε, γίνεται ακουστή άποψή τους. Επίσης, θα πρέπει να επικεντρώνεται στις πραγματικές προσδοκίες των πολιτών και να αναζητεί βιώσιμες πολιτικές λύσεις και συμβιβασμούς. Ε, με θεσμικές διαμάχες δεν πρόκειται να κερδίσουμε τίποτα. Με την αντιπαράθεση ε, ουτοπιών ή με την αναρχική συζήτηση που ακούγονται τα πάντα και τίποτα δεν υποφασίζεται, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Θέλουμε ε, μια ουσιαστική συζήτηση όπου τα θεσμικά όργανα, τα δημοκρατικά νομοποιημένα, μπορούν να λάβουν αποφάσεις και να κάνουν βήματα προς μια ε, ξεκάθαρη κατεύθυνση για μια πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική Ευρώπη που θα προσφέρει περισσότερη ευημερία στους πολίτες της. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάν για ένα λεπτό. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον της Ευρώπης, αγαπητοί συνάδελφοι. Σίγουρα θα συμφωνείτε με αυτό και θα το έχετε πει διάφορε φορέ στη προεκλογική εκστρατεία. Και τώρα μπορούμε να δείξουμε αν το εννοούμε πραγματικά. Γιατί η μελλοντική αυτή διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη είναι για διάσκεψη για το μέλλον τη επόμενη γενιά. Αυτή η νέα γενιά λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχει. Και ουσιαστικά περιμένουμε σεβασμό. Σεβασμό για του νέου που για τους πολίτες. Και αυτό έχουμε να το πούμε και στους πολίτες από το ECR που θέλουν να αποκλείσουν τη συμμετοχή των νέων με τις τροπολογίες τους. Από Αυτό περιμένουν όμως από το κοινοβουλίο μας και από, το... από τα εθνικά κοινοβούλια. Μόνο αν ε, συμμετέχουν οι νέοι πλήρω σε αυτή τη διάσκεψη θα δείξουμε ότι σεβόμαστε την άποψή τους και ότι μπορούν ενεργά οι ίδιοι να καθορίσουν το μέλλον τους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σα παρακαλώ, όχι σφαιρίγματα στην αίθουσα. Ο κύριο Μπούζελαγκρ για 1,5 λεπτό. Ακούγοντα τη συζήτηση αυτή, χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε ένα ισχυρό ψήφισμα εδώ στο Κοινοβούλιο που υποστηρίζει το μέλλον τη Ευρώπη. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία στοιχεία τα οποία α, ήδη ακούσαμε. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα. Και ακριβώ επειδή αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, προσπαθούμε να βρούμε λύσει και τα προβλήματα, όπως είπε ο κύριος Φερχόφστατ και η κυρία Ομπρέ, είναι όλες οι προκλήσεις της μετανάστευσης, κοινωνικών προτύπων κτλ. κτλ. Δεν μπορούμε να δώσουμε πλήρες απαντήσεις γιατί μας μπλοκάρουν σε ό,τι αφορά τις λύσεις που θέλουμε να δώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και κατά δεύτερον, τα εθνικά συμφέροντα. Ναι, επί του παρόντος θα πρέπει να προσπιστούμε τα δεν χρειάζεται να προσπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα, γιατί τα εθνικά συμφέροντα είναι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό. Η πλειοψηφία λοιπόν του Κοινοβουλίου είναι υπέρ του μέλλοντο και το μέλλον μπορεί να είναι μόνο ένα κοινό μέλλον για την Ευρώπη και αυτό σημαίνει να έχουμε ένα κοινό όραμα το οποίο θα μοιράζονται οι πολίτε. Και ελπίζω με την διάσκεψη αυτή να κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Ακριβώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο ε, για ένα λεπτό. Α, συγγνώμη. Κύριε Βελίμψκη. δεν σα είδα, ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Δέχεστε μπλε κάρτα. Έχετε το λόγο. Είναι για 30 δευτερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουζολάγκερ. Αναφέρατε ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ψήφισμα για το θέμα αυτό. Συμφωνώ. Να υπενθυμίσω όμω στο Κοινοβούλιο μια συζήτηση που θα κάνουμε για ένα πολύ έντονο ψήφισμα και για την Ουγγαρία και την Πολωνία. Εδώ δεν σημαίνει τίποτα. Πώς μπορούμε να αγγιηθούμε λοιπόν ότι το ψήφισμα που ψηφίζουμε τώρα δεν θα οδηγήσει σε κενά λόγια μόνο. Και να δούμε πραγματικά αποτελέσματα και το Κοινοβούλιο να μπορέσει πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα του. Ευχαριστώ. Απάντηση. Δύο στοιχεία για να μην είναι μόνο και ένα λόγια αυτά όπως είπατε. Καταρχάς, να υπάρξει συνέχεια σε ό,τι αφορά τα πορίσματα της συζήτηση, να γίνουν αλλαγέ στη διαδικασία, στη συνθήκη, να δούμε τον κανονισμό και τι ε, διαδικασίε που ακολουθούνται εδώ και στο Κοινοβούλιο και στα άλλα θεσμικά όργανα. Και κατά δεύτερον, να μην κοιτάξουμε μόνο τον bottom από κάτω προ τα πάνω, όπω είπε ο κ. Φερχόφστατ, αλλά και να πούμε στου πολιτέ ότι κοιτάξτε, αυτά είναι τα αποτελέσματα, συμφωνείτε ναι ή όχι. Μόνο με λογοδοσία θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τι πράξει μα. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μιλίμσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μιλάτε για το μέλλον τη Ευρώπη και θέλετε να το πάρετε στα χέρια σα. αλλά δεν καταφέρετε καν να πάρετε στα χέρια σα το παρόν τη Ευρώπη και τα σημερινά προβλήματα, τη μετανάστευση. Ούτε αυτά είναι σε θέση, Όπω και τη φύλαξη των ιστορικών συνόρων. Ούτε και αυτό μπορείτε να το ε, ε, πετύχετε διατήρηση της οικονομίας ύστερα. Έχουμε μια πολιτική μηδενικών επιτοκίων, αρνητικών επιτοκίων, ασθενής η οικονομία και δεν μπορούμε να τα βελτιώσουμε αυτά. Η κρίση του κλίματος, εδώ υπάρχει κάποια άμα, πρόοδος, αλλά εδώ και πάλι χρησιμοποιείται την πολιτική για να πάρετε λεφτά από τα τσέπη του κοσμάκη και θα αποτύχει και πάλι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάθε μήνα έχουμε 120 χιλιάδες οχήματα τα οποία φεύγουν από το τις Βρυξέλλες να έρθουν στο Στρασβούργο. Πώς λοιπόν συνάδουν όλα αυτά. Να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν τα προβλήματα. Τα εθνικά μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους μόνα τους. Και εδώ είναι το επιτυχές και ε, καλό μέλλον για την Ευρώπη. Κύριε Βιλίμς, έχετε, μία μπλε κάρτα από την κυρία Ντέμα. Μπορείτε να τη δεχτείτε. Παρακαλώ. Υποβάλλετε την ερώτησή σας. Κύριε Βιλίμσκι, δεν μιλήσατε καθόλου επί της ουσίας. Να σας ρωτήσω όμως, γιατί είσαστε αντίθετοι να συμμετέχουν οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάσκεψη, να κάνουν ανταλλαγή απόψεων, να μα πούν αυτοί ποια είναι το όραμά του για το ε, μέλλον τη Ευρώπη. Αν αντιστεκόμαστε και δεν θέλουμε να ακούμε την ε, άποψή του, τι νόημα υπάρχει απάντηση. Εκτιμώ ιδιαίτερα το άτομό σα, αλλά είστε καινούργια εδώ στο Κοινοβούλιο. Ήμουν εδώ και την προηγούμενη θητεία και έχω πιστοποιήσει όλα αυτά που έχουν ζητηθεί τόσες πολλές φορές για το μέλλον τη Ευρώπη με τη συμμετοχή των πολιτών, των ομάδων, συμφερόντων κτλ. Δεν υπάρχει καμία συνένεση και το Κοινοβούλιο δεν τολμά να δώσει κατεύθυνση. Μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης τόσες πολλές φορές και ε, ως σήμερα το Κοινοβούλιο δεν έχει κάνει οποιαδήποτε διαπίστωση. Αυτό και κατηγορώ. Αυτή είναι η κατηγορία μου το Κοινοβούλιο. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Μπουσαντέ, Κύριε Πρόεδρε, Δέκα χρόνια μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και μετά από μια χρηματοπιστωτική κρίση, μια μεταναστευτική κρίση και το Brexit, δεν έχουμε λύσει ακόμα ε, κανένα από αυτά τα προβλήματα. Καλό είναι που συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης, ε, αλλά από ό,τι φαίνεται η λύση είναι να προχωρούμε προς την ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης που στην ουσία μας οδηγεί προς τον κρεμό, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία μας έφερε εδώ που είμαστε. Εμείς θέλουμε μια ελεύθερη διάσκεψη, ναι, ε, που όμως να μην αποκλειστεί η άποψη του 20% ε, των πολιτών ε, και των βουλευτών που αποκλείστηκαν από, την, από το ψήφισμα. Τα κράτη-μέλη δεν είναι δυνατόν να και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να αποκλείει το 20% των πολιτών της Ευρώπης. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που θα αποτελείται από ελεύθερα κράτη, από από κυρίαρχα κράτη και να σας θυμίσω κάτι που ξεχνάτε το μέλλον περνάει από τις παραδόσεις και από την χριστιανική μας ε, παράδοση και την ιστορία μας. Ε, έχετε έτοιμα για ε, μπλε κάρτα, κύριε Μπουξαδέ, το δέχεστε. Έχετε, υπάρχει μια ερώτηση για σας, τη δέχεστε. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να αποτρέψω τη δημιουργία ενός μύθου, γιατί δύο μέλη της ομάδας σας ε, πήραν το λόγο και λέτε ότι εξαιρείστε και αποκλείστε από την κατάρτιση του ψηφίσματος αυτός. Αυτό δεν στέκει. Δεν ξέρετε ότι η δική σας επιθυμία ήταν. Εσείς αποσυρθήκατε. Όλοι οι υπόλοιποι στεναχωρέθηκαν, λυπήθηκαν. Θα θέλαμε να υπάρχει ένα ψήφισμα από όλες τις πολιτικές ομάδες. Εσείς αποσυρθήκατε. Εμείς δεν σας κλείσαμε απ' έξω. Το γνωρίζετε αυτό.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 Λυπούμε που σας ακούω να το λέτε αυτό. Είμαι και εγώ μέλος της ε, ΑΦΚΟ ε, και ε, ήδη από την πρώτη συνεδρίαση μας παρουσιάστηκε ένα ψήφισμα που είχε υπογραφεί από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες και από εκεί και πέρα είπατε να υποβληθούν τροπολογίες, αλλά ούτως ή άλλως ήταν ήδη γραμμένο το έγγραφο. Εμείς πιστεύω ότι θα έπρεπε να δουλέψουμε από την αρχή και με σεβασμό προς τους πολίτες μας, όλους τους πολίτες. Ο για να γίνει η Ενωμένη Ευρώπη πιο ελκυστική και πιο ισχυρή, χρειάζεται να γίνει πιο δημοκρατική, πιο κοινωνική, πιο οικολογική και πιο δίκαιη. Μόνο έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο της οπισθοδρόμησης και της επιστροφής σε ένα μαύρο παρελθόν που επιδιώκουν ανοιχτά πια οι δυνάμεις της αντιευρωπαϊκής λαϊκίστικης ακροδεξιάς. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει ο διάλογος αυτός να γίνει με ισχυρό το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου όχι μόνο μεταξύ των ελίτ αλλά κυρίως με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική μου ομάδα της αριστεράς συνυπογράφει αυτό το ψήφισμα παρότι θα το θέλαμε ριζοσπαστικότερο και μας εντυπωσιάζει η απόλυτη άρνηση της άκρας δεξιάς όχι μόνο να στηρίξουν αυτό το ψήφισμα αλλά και η άρνησή τους να δεχθούν τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτό το διάλογο. γιατί φοβόσαστε τη συμμετοχή των πολιτών; Ευχαριστώ κύριο Σίντζιτς. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, φυσικά έθνη και κράτη υπήρχαν και πριν την την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη θα υπάρχει και μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αναγνώρισης της Κροατικής Δημοκρατίας. Και μάλιστα εγώ άκουσα τους διάπειρους υπέρμαχους Ευρώπης που επιτέλους παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος. Αυτό είναι για μένα επιβράβευση προσωπική. Ε, μπράβο, μπράβο που αναγνωρίσατε τα σφάλματά σας. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα για να βρεθούν λύσει. Ε, θέλουμε, σολιδε... Ε, θέλουμε αλληλεγγύη. Όταν ε, έχουμε πλημμύρες στη Σλοβενία, αμέσω σπέβδουμε να βοηθήσουμε τη Σλοβενία ή όταν έχουμε πυρκαγιές αλλού, αμέσω σπέβδουμε να βοηθήσουμε. Αλλά πού είναι η αλληλεγγύη προς την Κροατία. Την αλληλεγγύη την καταπατήσατε με τις περιοριστικές σας πολιτικές. Τώρα θέλετε εξωθείτε την Κροατία να μπει στην Ευρωζώνη. Ε, βέβαια θα χάσουμε έτσι πολλούς μηχανισμούς για να ξεφύγουμε από την κρίση, όπως είναι ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τι θα κάνουμε, θα χάσουμε όπως η Ελλάδα το 25% του ΑΕΠ μας αν μπούμε στο Ευρώπη. Ε, θέλετε να μας εξολοθρέψετε, γι' αυτό θέλετε να μας βάλετε στο ευρώ. Η κυρία Χιούμπνερ για 1,5 λεπτό. Συνάδελφοι, αυτή η διάσκεψη δύο ετών μπορεί να αποτελέσει κάτι διαφορετικό πέρα από ότι αυτό που φαντάζονται οι λαϊκιστέ πολιτικές. Έχουμε μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια ε, συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Μπορεί να είναι μια συζήτηση μεταξύ ε, ίσων σε ό,τι αφορά το διάλογο που πρέπει να γίνει για το μέλλον της Ευρώπης και η διάσκεψη αυτή αποτελεί μια πολιτική διαδικασία και μπορεί να έχει ε, την δική της προστιθέμενη αξία, να ανανεώσει την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, να προωθήσει την ενότητα της Ένωσης και την εθαγένεια και το αίσθημα ιδιοκτησίας μεταξύ των πολιτών. Ένας τέτοιος ανοιχτός διάλογος μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτυχθεί με αμοιβαιότητα προς τους πολίτες και πιστεύω ότι η διάσκεψη αυτή αποτελεί μια συνέχεια σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι εκλογές του 2019 δημιούργησαν μια κοινή ε, ευρωπαϊκή αφήγηση και όχι τόσο πολύ 28 ε, διαφορετικές ε, ιστορίες. Αυτές οι εκλογές απέδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν πιο πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το παρελθόν. Ξέρουμε ότι θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί να μιλήσουν για την επανακοσμιοποίηση, το κλίμα, την μετανάστευση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανταγωνιστικότητα, την ψηφιοποίηση και όλα αυτά. Θέλουν να συμμετέχουν λοιπόν οι πολίτες και να δώσουν απάντηση στις προκλήσεις σύμφωνα και με τα όνειρά τους και με τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να αντράξουμε την ευκαιρία για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Χούμπνερ, υπάρχει μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Όχι, δεν δέχομαι. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε την συζήτηση. Ωραία, προχωράμε λοιπόν στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Γκραπίνη. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλθε ε, μεγάλη κρίση και επομένως θα πρέπει να συζητήσουμε ε, για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να συζητήσουμε και με τους πολίτες παρότι εμείς ήδη είμαστε μέλη της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και εκπροσωπούμε τους πολίτες και μπορούμε να μιλήσουμε εξ ονόματός τους αλλά βεβαίως εάν ένα μέτρο αποτύχει ή δεν είναι αρκετό πρέπει κανείς να προστρέξει και σε άλλα μέτρα. Είναι σημαντικό να ενταχθεί αυτή ε, η διάσκεψη, αυτή η νέα πλατφόρμα ε, με τρόπο ώστε να ε, έρθουν πιο κοντά οι πολίτες με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι σημαντικό επίσης ε, είναι να μην αυξήσουμε το κόστος ε, και την γραφειοκρατία και να προχωρήσουμε στην αποτελεσματικότητα. Ε, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η επικοινωνία μας με τους πολίτες. Ευχαριστώ ένα λεπτό ο κύριος Γκιόρενς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα της διάσκεψης, η διάσκεψη η ίδια θα είναι δύσκολη, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην ξεκινήσει. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε όλοι μαζί, γιατί ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε μέχρι τώρα και λειτουργούμε θα μας ρίξει στη δεύτερη κατηγορία. Ε, θα πρέπει να αναλύσουμε ε, τον, τους λόγους ε, της παράλυσης μας. Θα πρέπει να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον θα μπορέσουμε να δώσουμε φωνή στους νέους και στους πολίτες. Και γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι ε, θα πρέπει να δούμε λίγο και τα μηνύματα των νέων Βρετανών που αντιτίθεται στο Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Μπρέγερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, πώς θα καταφέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει πολιτικές απαντήσεις για την πλειοψηφία των πολιτών και όχι για τους, πολιτικούς, και όχι για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Πώς μπορούν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους οι πολίτες με άμεση δημοκρατία για να κερδίσουμε το, την εμπιστοσύνη των πολιτών σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό έργο. Για να προστατεύσουμε την Ευρώπη από τους εθνικιστές. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε λοιπόν μια βάθρον ανάλυση της Ευρώπης. Αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ελπίζουμε ότι θα δώσει κάποιες απαντήσεις και κάποιες μικρές βελτιώσεις. Αλλά το να περιμένουμε ε, από τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων να μεταρρυθμίσουν τα θεσμικά όργανα αυτά είναι ένα προβληματικό στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία κατευθείαν άμεσα άμεση διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή των πολιτών με μία δημοψήφισμα να αποφασίσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν να έχουν. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Μπαρτέλα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. η κοινωνική Ευρώπη που θα προστατεύει πιο δημοκρατική θα τα ακούμε εδώ και 30 χρόνια. Ε, την ίδια υποδό ακούμε από τους πολιτικούς ηθήνοντες, αλλά είναι φρούδες υποσχέσεις που δεν τηρούνται. Κανένα θεμητό και βιώσιμο σχέδιο για την Ευρώπη δεν θα δει το φως της ημέρας αν δεν στηρίζεται σε ελεύθερη συνεργασία μεταξύ των εθνών και τη σεβασμό της κυριαρχίας του κάθε κράτους. Δεν είναι επιλήψη με μόνο στη δομή της Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως ε, είναι ε, αξιόμεμπτη η πολιτική της. Γιατί ε, έχουμε τεχνητή τη νοημοσύνη, τεχνολογικές εξελίξεις, προστασία του κλίματος, ε, του περιβάλλοντος, αλλά έχει αποτύχει η Ευρώπη σε όλα αυτά. Θα πρέπει να ανταγωνιστούμε την Αμερική, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία. Στην ουσία όμως είμαστε ανήμποροι. Έχω μια ευχή. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, να είναι ευκαιρία για μια αλλαγή, ριζική αλλαγή πορείας. Αλλά δυστυχώς δεν έχω ψευδεστήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαρντελά, ο κύριος Χαμπίμπ θέλει να σας θέσει ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Τη δέχεστε? Μάλιστα. Ο κύριος Χαμπίμπ, ευχαριστώ. Κύριε Μπαρντελά, συμφωνείτε μαζί μου ότι το, ο τίτλος ε, της διάσκεψης είναι παραπλανητικός. Θα έπρεπε να είναι διάσκεψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Συμφωνείτε ότι δεν χρειάζεται καν διάσκεψη γιατί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μάλλον σκοτεινό και πολύ πιθανό να διαλυθεί σχετικά σύντομα. Εγώ δεν συγχαιώ την Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που εφήβρε την έννοια του έθνους ε, και περιλαμβάνει από τα αρχαιότερα έθνη του κόσμου. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο έχει να καταστρέψει τα έθνη και είναι ένα σχετικά νέο δημιούργημα και χαίρομαι που ο Βρετανικό λάο θα ανακτήσει την ελευθερία του. Πάντως δεν μπορούμε να φανταστούμε ευρωπαϊκή συνεργασία χωρίς την ε, ισχύ της μεγάλη Βρετανία. και θα πρέπει να βρούμε ένα νέο, μια νέα μορφή ε, ευρωπαϊκής ε, συνεργασίας μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να διευκολύνω τη συζήτηση θα συνεχίσω να δίνω ερωτήσει με μπλε κάρτα, αλλά μόνο σε έναν ομιλητή, Άννα. Ε, θέμα. Ο κύριος Τσίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν οι πολίτες ε, διαπιστώσουν ότι παρά τη νέα πράσινη συμφωνία έχουμε ε, ε διατάξεις που υποχρεώνουν τα φορτηγά να κυκλοφορούν κενά στην Ευρώπη σε ταξίδια επιστροφής, τότε θα δυσαρεστηθούν. Επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε προτάσεις για άμυνα και να μειώνουμε τον προϋπολογισμό συνοχής της πολιτικής συνοχής, κάτι που θα φέρει σε ακόμη πιο δινή θέση τις ε, μειονεκτούσες περιοχές της Ένωσης και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δεν θέλουν αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν ζητούν περισσότερη Ευρώπη. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει μόνο οι μεγάλες χώρες να εκπροσωπούν τη θέση τη Ευρώπης. Δεν είναι μόνο οι ισχυρέ χώρες η φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα δυσαρεστεί και πάλι του πολίτε. Επίσης, αν έχουμε υπερεθνικά ψηφοδέλτια, ούτε αυτό θα τους ικανοποιήσει. Έτσι, κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε τα πλεονεκτήματα τη Ευρώπη. Όποιο θέλει τα πολλά, μερικέ φορέ χάνει και τα λίγα. E η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει τις πολυεθνικές εταιρείες, διευκολύνει τους πλούσιους και τους ισχυρούς. Και αυτό το είδαμε ε, για το κλίμα, το περιβάλλον, τη, τα κοινωνικά δικαιώματα. Θέλουμε μια πιο ισορροπημένη συνεργασία όπου οι πολίτες, η φύση και το κλίμα θα βρεθούν στο επίκεντρο. Θέλουμε λοιπόν μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό που δεν θέλουμε είναι μια προκαθορισμένη συζήτηση όπου το αποτέλεσμά της είναι περισσότερη συγκέντρωση και πιο απορριθμισμένες αγορές. Θέλουμε μία ανοιχτή και πραγματική συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων. Είμαστε δηλαδή υπέρ του ψηφίσματος, αλλά δεν ε, φοβόμαστε ποτέ να βοηθήσουμε, να ζητήσουμε τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών. Και σας προειδοποιώ, αν δεν έχουμε ε, γνήσια ανάμειξη των πολιτών και ευρύ ανάμειξη των πολιτών, οι πολίτες δεν πρόκειται να μας συγχωρήσουν. Κύριε για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το μέλλον των Ηνωμένων Βασιλείου είναι λαμπρό γεμάτο με ευκαιρίε. Γιατί έχουμε την πολιτική βεβαιότητα ότι θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο εβδομάδε μόλι. Η ευκαιρία να μπορέσουμε λοιπόν να αποφασίσουμε για τη χώρα μας όπως θέλουμε, όχι όπως μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ευκαιρία να είμαστε μια χώρα υψηλής ανάπτυξης, χαμηλής φορολόγησης, φύση τεχνολογίας που θα συναγωνίζεται με τα άλλα κράτη χωρίς γραφειοκρατία και προστατευτισμό περιττό. Να έχουμε λοιπόν μια σωστή πολιτική μετανάστευση που θα λειτουργήσει για την οικονομία μας, για τον λαό μας. Την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε κρατικές επιδοτήσεις ε, για τις στρατηγικές μας ε, επιχειρήσεις. Τα ποσοστά απασχόλησης είναι σε ποσοστά ρεκόρ ε, και το ίδιο ισχύει για την αργία που είναι εξίσου σε ποσοστό ρεκόρ χαμηλή. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους μας. Σας συστήνω λοιπόν την ευκαιρία θα πρέπει το μέλλον να είναι λαμπρό και για τις υπόλοιπες 27 χώρες αν ακολουθήσετε το παράδειγμά μας και μειώσετε τον έλεγχο. Ο κύριος Κάρας για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι, συμφωνούμε στην πλειοψηφία μας ότι το μέλλον μας θέλει μια πιο αξιόπιστη και πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε εμείς όλοι, οι πολίτες ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, των ε, περιφερειών, θα πρέπει λοιπόν το μέλλον να είναι φίλος μας. Θα πρέπει φίλος μας και σύμμαχοι μας να είναι και πολίτες. Το μέλλον της Ευρώπης και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο προσκήνιο θα πρέπει να μπει πάνω από τα όρια των κομμάτων. Το μέλλον χρειάζεται ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας να σταματήσει η διαδικασία ε, ομοφωνίας ε, στην λήψη αποφάσεων, το δικαίωμα σε το θέμα της καταορισμού του προπολογισμού. Το μέλλον χρειάζεται μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που θα είναι καθοριστική για τη μεγάλη αυτή του κόσμου και πέρα από την πολιτική, θα, θα ορίζει και την πολιτική, την εξωτερική και την πολιτική άμυνα. Το μέλλον μας λοιπόν προαπαιτεί ευρωπαϊκές ε, απαντήσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Μια ιστορική αγορά χωρί ε, σύνορα. Το μέλλον μας χρειάζεται έναν προπολογισμό που θα ανταπεξέλθει στο ύψο των προκλήσεων όλη τη Ευρώπη, που θα επενδύσει στο μέλλον και ως εκ τούτου σας λέω ότι το μέλλον προαπαιτεί διάλογο, ευρωπαϊκή συνείδηση, κοινή δράση. Εμείς ως κοινοβούλιο θα πρέπει να τα διαθέσουμε όλα αυτά με τα ένα εκατομμύριο επισκέπτες μας, με την υψηλή προσέλευση στις κάλπες και με τα ε, γραφεία σύνδεσης. Κύριε Καράς, λέει η Πρόεδρος και διακόπτη. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Πιζαπία. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε κυρία Πρόεδρε. Πέρασαν περίπου 80 χρόνια από την εποχή που ο Αλτιέρο ε, Σπινέλη και ο Ρώση ε, αποκλεισμένοι ε, σε, από το καθεστώς το φασιστικό έγραφαν σε μια επιστολή τους χρειαζόμαστε ανανέωση και συμπερίληψη. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης μας δίνει μια εξαιρετική, ίσως μάλιστα την τελευταία ευκαιρία για αλλαγή και συμμετοχή. Όχι μονάχα στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στις περιφέρειες και οι ε, ε, στην Ήπεθρο ε, και ακούγοντας και την άποψη όσων δεν συμμερίζονται το παρόν σύστημα. Χρειαζόμαστε ένα, μια δομή η οποία θα είναι σε θέση να ε, τροποποιήσει, να μετατρέψει τις ε, ε, ιδέες και τα λόγια σε μέτρα και πράξεις, γιατί διαφορετικά θα σπαταλήσουμε μία από τις τελευταίες ευκαιρίες αλλαγής και σίγουρα αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ και θα οπισθοδρομήσει και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία προς τα εμπρός, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε δεν είναι ούτε εύκολος ούτε σίγουρος, αλλά θα τον ακολουθήσουμε με πεποίθηση και στένωση. Η κυρία Χαραντζόβα. Ε, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα καθορίσει ε, το κοινό μας μέλλον. Ε, οι ίδιοι οι πολίτες ε, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ε, να εκφραστούν. Γι' αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι παρόντες στην διάσκεψη αυτή για το μέλλον της Ευρώπης. Ακούμε τις ε, εκκλήσεις τους εδώ και χρόνια. Τώρα όμως θα πρέπει να ακούσουμε και τις επικρίσεις τους. Πρέπει να τις ακούσουμε, να τις κατανοήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα. Υπάρχει αυτή η φούσκα των Βρυξελών, αυτή αυτός ο πύργος της Βαβέλ των Βρυξελών ε, που δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ότι γύρω του ο κόσμος αλλάζει. Θα πρέπει να ε, δώσουμε απαντήσεις. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κοφεύσουμε ε, και να αποστρέψουμε το βλέμμα από τις ανάγκες των πολιτών. Κυρία Χαραντζόβα, υπάρχει μία μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Παρακαλώ, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Κυρία ε, Χαραντζόβα, ε, χαίρομαι που αναφερθήκατε σε ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών. Εσείς πώς θα βλέπατε αυτήν την συμμετοχή των πολιτών, πώς θα μπορούσατε να οργανώσετε αυτή τη συμμετοχή. Εύκολη είναι η ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, εάν αποφάσιζα εγώ, θα έλεγα ότι μονάχα νέοι και μονάχα πολίτες θα έπρεπε να συμμετέχουν. Ε, όταν, έρχομαι, όταν πηγαίνω στην περιφέρεια της Εθνικής Δημοκρατίας, μιλάω με τους νέους, μιλάω με τους πολίτες ε, και πραγματικά ε, πρέπει να τους ακούσουμε όλοι, όλοι, στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριο Σέντσλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Brexit θα πρέπει να είναι προειδοποίηση για όλους μας για το τι συμβαίνει όταν ο κοινός θνητός βλέπει ως απόμακρη, ε, ανέθινη ε, την Ευρώπη και γίνεται θύμα ε, ακροδεξιών δημοκόπων που στρέφουν τον κόσμο εις, βάρο, εις Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζωπυρώνοντας τον ευρωσκεπτικιστικό φόβο. Είναι πια αργά για το Ευρωπαϊκό ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο το κακό έγινε. Αλλά θα πρέπει να είναι το πάθημα αυτό δίδαγμα για όλους μας. Και αν ε, θα έχει κάποιο νόημα ε, η διάσκεψη, θα πρέπει να ακούσει και να φογκραστεί τους πολίτες. Δεν θα μπορεί να περιοριστούμε σε μια τυπική διαδικασία που απλώς θα επιθυμούμε τη σφραγίδα των πολιτών. Θα πρέπει να επηρεάσει πολιτική, να επηρεαστεί η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην φημωθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και οι πολίτε όπω συχνά συμβαίνει. Αυτή η ζωτική σημασία διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να ζητήσει τη γνώμη όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και εμεί ω φιλοευρωπαίοι πιστεύουμε να... και θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία και είμαστε υπερήφανοι για αυτή την δυνατότητα που μας δίνετε. Ευχαριστώ. Κυρία Χώτης Αρίστη, επόμενη ομιλήτρια και ζητήσετε προηγουμένως διαδικασία μπλε κάρτας. Δεν θα στο επιστρέψω γιατί ο χρόνος πιέζει και οι σύμβουλοι μου συνιστούν να μην δίνω πια το λόγο για ερωτήσεις με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Στις 12 έχουμε πανηγυρική συνεδρίαση και θα πρέπει να ετοιμάσουμε την αίθουσα. Οπότε δεχτείτε την απόφαση μου τώρα. Τα διαδικαστικά μπορούμε να τα συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Η κυρία Χουτεσάρη για ένα λεπτό. Συγγνώμη, μια στιγμή κυρία Χουτεσάρη. Ένα διαδικαστικό προηγουμένως. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε αλλά διαφωνώ με την απόφασή σας για τις μπλε κάρτες. Μία ώρα θα έχουμε μεταξύ του τέλους της συζήτησης αυτής και την έναρξη της επόμενης συζήτησης. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να, το συζητή, ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος. Θα σας παρότερη να συνεχίσουμε τη συζήτηση και με μπλε κάρτες, γιατί πραγματικά αναζωογονήθηκε η συζήτηση χάρη στις μπλε κάρτες. Αμφισβητώ λοιπόν και διαφωνώ με την απόφασή σας να τις διακόψετε. Θα σας παρότεινα και θα σας ενθάρρυνα να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή και τις μπλε κάρτες. Έχω... λατρεύω τις μπλε κάρτες και το σύστημα και δουλεύει, αλλά έχουμε μείνει πίσω στο χρόνο και αν συνεχίσουμε τη ζήτηση με μπλε κάρτες δεν θα έχουμε καιρό στην πανηγυρική συνεδρίαση. Πολύ ευχαρίστως αργότερα να συζητήσουμε πώς ε, στο μέλλον θα χειριστούμε τη διαδικασία αυτή. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Παρακαλώ δεχτείτε την απόφασή μου και θα λάβω τα σχόλιά σας. Ίσως στο μέλλον χρειαστούν κάποιες αλλαγές στη διαδικασία. Κυρία Χουτεσάρη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα η συνεργασία είναι εννοητή μόνο με τους ομοειδεάτες, μόνο με όσους συμφωνούν. Και αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει και εδώ. Όσοι έχουν αντίθετη γνώμη παραμερίζονται. Θεωρείται την αντίθετη γνώμη ως απειλή. Και τον εθνικισμό και τον Brexit ε, το θεωρείται επίσης απειλές. Και εμείς σας θεωρούμε απειλές για τη κυριαρχία των εθνών κρατών. Επίσης, ε, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικοί θύνοντες θεωρούν ότι θα πρέπει για μία ακόμη φορά να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν το σοσιαλισμό. Ε, το Brexit τους πανικόβαλε. Και μάλιστα αφαιρέθηκαν και τα σημαίακια από τα έδρανά μας. Λέτε ότι θέλετε να εμπλακούν οι πολίτες στην όλη διαδικασία αλλά Θέλετε τελικά μόνο τους ομοειδεάτες σας να εμπλέξετε. Γιατί δεν εμπλέκετε τους λαϊκιστές στη συζήτηση, αλλά μόνο τους πολίτες. Και για αυτούς που παρακολουθούν το ρολόι, δώσαμε 30 δεύτερα. Δεν ξεπέρασε το χρόνο τα ε, η ομιλητρία. Ο κύριο Έπιγκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Όντω είναι σε σταυροδρόμι η Ευρώπη, κυρίε και κύριοι. Το ψήφισμα της πλειοψηφίας είναι σαφές. Θέλετε μια, ένα επικυριαρχό ευρωπαϊκό κράτος με το στρατό του, με τη δική πολιτική και να κάνετε επαρχίες στα κράτη-μέλη. Οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί έχουν διαφορετικό όραμα για την Ευρώπη. Μια κοινότητα ε, επικυρίαρχων κρατών, μια συνεργασία μεταξύ κρατών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πιο πολύ ε, εξουσία στα κράτη και να μειωθεί η βαριά γραφειοκρατία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν μια παράλληλη διαδικασία με ανταγωνιστικό έργο. Θα στραφούμε στα κρατημέλη και θα κάνουμε συζήτηση μετά με τους ε, πολίτες και θεωρούμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφανθούν σε δημοψηφίσματα. Να ρωτήσουμε λοιπόν τους πολίτες, όχι μόνο ομικείο κτλ και πολίτε σε διάφορε περίεργε θέσει. Όχι, να ρωτήσουμε άμεσα του πολίτε για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή ε, της Ευρωπαϊκής και όχι μόνο επιδοτούμενες οργανώσεις. Ευχαριστώ, κυρία Φόξ, για ένα λεπτό. Είναι η καλύτερη συζήτηση αυτή που έχω ακούσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Πολύ καλή Προεδρία, κυρία Μακίνες. Έχουμε ακούσει κάποιες ε, ειλικρινές, απόψει. και ο κ. Φαρχόφστα τα έχει δείξει τα πνεοφροσύνη και να γνωρίζει ότι έχουμε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Όλε αυτέ οι διαβουλεύσει έχουν ένα εξή κίνδυνο, ότι επιφανειακά θα υπάρχει συμμετοχή του πολίτη, αλλά ουσιαστικά είναι στυλιζαρισμένε και στημένε συζητήσει. Οι πολίτε κάνουν συζήτηση διαρκώς ελεύθερα, χωρίς τη βοήθεια των γραφειοκρατών. Οι γραφειοκράτε φωνάζουν τις απόψεις τους ε, στις εκλογές, στα δημοψηφίσματα, αλλά τους απορρίπτει ο κόσμος. Όταν ε, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρίνουν ε, την πολιτική λιτότητα στα θεσμικά όργανα, πολλοί ε, στα πολιτικές, πολιτικές ομάδες κοφεύουν. Είστε ε, λαϊκιστές, είστε ακροδεξιά, κατηγορούν. Χειραγωγείτε, λένε στους εκλογείς. Με, άλλες, ε, με άλλα λόγια, δεν μπορείτε να ακούσετε τους πολίτες αν δαιμονοποιείτε τους πολίτες αυτούς και κάνετε στη συνέχεια τα πτή η πρόεδρος στο σημείο αυτό. Δεν σας ακούει κανείς, αλλά συνεχίστε άμα θέλετε να μιλάτε μόνοι σας. Δεν έχετε μικρόφωνο πλέον γιατί ξεπεράσατε το χρόνο ομιλία σας. Ο κύριος ε,